Καλημέρα. Αρχή η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, ε, παραμονές του Πάσχα. Καλωσορίζω του αραλέου και του Γενναίου που ήρθαν. Κανονικά ε, είχαμε και το απόγευμα συνεδρίαση, αλλά δεν μπορέσαμε να γεμίσουμε την ημερήσια διάταξη, γιατί κανένας δεν ήταν πρόθυμος να βάλει θέμα το απόγευμα, οπότε και ε, καταργήθηκε. Έχουμε την ημερήσια διάταξη, δεν έχει ζητήσει κανεί αλλαγή. Δεύτερον, ε, ανακοινώσει της Προέδρου. Ε, σας παραπέμπω στο Cont News, θα δείτε τις γλώσσες που έχουμε. Και σε ένα τέταρτο ε, θα έχουμε μια ώρα ακρόαση με την υποψήφια της Ουγγαρίας για το ελεκτικό συνέδριο και θα έχουμε και ανάγκη για απαρτία. Μετά έχουμε την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και θα συζητήσουμε τα δύο ταξίδια μας, δύο αποστολές, Ιορδανία, ε, Λίβανο και Τουρκία. Και θα ασχοληθούμε και με την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παγκόσμιας Τράπεζας στην Περισσινή που προκάλεσε κάποιο άλλο και κάποια <laughs> προσοχή. Ερχόμαστε στο σημείο 3 της ημερής της διάταξης, ε, εκτέλεση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι γνωμοδότηση αυτή, Συγητής ο συνάδελφος Τάκουλα. Θέλετε το λόγο κύριε Τάκουλα. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι μπορώ να είμαι σύντομο, να ευχαριστήσω μόνο τους και για τη συνεισφορά τους κατά την εκπόραση της νομοδότησης αυτής και νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε έτσι σε ένα καλό πνεύμα και κλίμα. Μάλιστα, αρχίζουμε. Τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αυτό θέλει έλεγχο μας, τροπολογία 3, ηλεκτρονική επαλήθευση. Για να δούμε πώς έχουν οι πλειοψηφίες εδώ και οι συσχετισμοί. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμό 4 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμό 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο. Παρακαλώ η τροπολογία 13 ηλεκτρονικά. Από το ΕΛΚΑ υπάρχει ένας υπεράριθμος ψηφίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία περιθών 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 καταπίπτει, 17 επίσης, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 20 καταπίπτει, 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 It is rejected. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Against abstentions. Κατά αποχές. 32 υπέρ. Τώρα δεν ψηφίσαμε. Κατά αποχές. Α, ας την επαληθεύσουμε παρακαλώ την 32. Check this over. Εγκρίνεται. 33. Καταπίπτει. Συμβαστική 1. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 36 Υπέ. Κατά. Αποχές. Ας την επαληθεύσουμε παρακαλώ αυτή. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά για καλό και για κακό. Πάλι περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Πέρας. Απερίφθεντος. 37. Καταπίπτει. 38 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42. Ορίστε. Έλεγχος για τη 41, μάλιστα. Θα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασα. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 καταπίπτει. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές Μπορώ να δω ξανά ε, τους κατά παρακαλώ. 45. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ, κατά αποχές Ας το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ, την 56 πολυθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, δηλαδή απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Ας την ελέγξουμε παρακαλώ την 60. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρινέται. 66 υπέρ. Κατά αποχές. Μπορούμε να την ελέγξουμε παρακαλώ την 66 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίφθη. 67 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται 68 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται 69 είπε. Κατά αποχές 69. Για την ελέγξουμε αυτή παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Mm. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο τώρα της γνωμοδότησης ονομαστικά αρχίζει ψηφοφορία. The vote is closed. 19 ψήφοι υπέρ, 2 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Τάκουλάμ. Η επόμενη ψηφοφορία. Μαζί Παράταση κυρίω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, θέσπιση τεχνικών και τα λοιπά. Θέλετε το λόγο, ναι, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συνδέλφου ε, και ιδίω του Σκιώδη ε, που συμμετείχαν στην διαδικασία αυτή. Είχαμε πολύ οικοδομητικέ συζητήσει και νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία σε ό,τι αφορά το ΕΦΣΙ. Ωραία, λέει και η πρόεδρο. Ξεκινάμε με τροπολογία 12. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήταν ταυτόσημη με 16 και 17 όχι εγκρίθηκε ναι με συγχωρείτε συγγνώμη εγκρίνεται οι 15 μέχρι 17 είναι ταυτόσιμα, άρα εγκρίνονται όλα. 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ, 19 Ελέγχουμε την 20, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε, την 20. Check is over. And it is adopted. Εγκρίνεται. 20-21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 και 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι να ελέγξουμε ελέγχουμε την 27 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται σαφώς συγγνώμη δεν το κατάλαβα 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. Ή καλύτερα να ελέγξουν παρακαλώ. Την 29. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολία 30 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήταν 34 ταυτόσιμο πάμε στις 36 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε παρακαλώ από κοινού τις 36 35 όχι Α, είναι ασύμβατη. Την 36 τότε να ελέγξουμε. Την 36 παρακαλώ, έρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 35 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ και την 35. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε πράγματι. 37 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 καταπίπτει. 41 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ 43 τροπολογία άρχιτη ψηφοφορία πέρασε απορρίφθηκε 44 ψήφι περ κατά αποχές απορρίπτεται 46 κατά τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι περ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται το ελέγχουμε όμως το πρώτο τμήμα της 46 παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτεται με την ίδια διαφορά ψήφων. 47 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίφθηκε. 48 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίθηκε. 49 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίφθηκε. 50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 πλένα υπέρ κατά αποχές Προπολογίε τροπολογίες 54-55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 56 και 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 58 και 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 60 υπέρ κατά να ελέγξουμε να ελέγξουμε την 60. Φέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 61 και 62. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 είναι τεχνική φύσεως 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε την 69 ναι άρχεται η ψηφοφορία ένας υπεράριθμος ε, στο ΕΛΚ παραπάνω. Όχι. Εντάξει. Συγγνώμη. Είμαστε εντάξει. Την 69 ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Τροπολογία 5 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά απόχέ, απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχέ. απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά απορρίπτεται 86 υπέρ κατά απορρίπτεται 87 υπέρ κατά απορρίπτεται 88 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται 90 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 υπέρ κατά εγκρίνεται 91 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 92 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 93. Let's check 93. Check is over. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 95 κατά καταπίπτει. 96 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συγγνώμη, 102 ήταν αυτή. 103 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 140 αποκρύπτεται, μάλλον 104 ηλεκτρονικά νομίζω εγκρίνεται. 104, Έλεγχος 104 ολοκληρώθηκε, απορρίφθηκε 104. 105 υπέρ, κατά αποχές, απορρίφθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότης. Ονομαστικά έχετε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 18 προς 4. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Και τώρα περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη με συγχωρείτε τον κύριο Τάραντ. Δεν ξέρω, θέλετε το λόγο κύριε Τάραντ. Όχι, Πρόεδρε, α ψηφίσουμε, λέει ο κύριο Τάραντ. Ε, εντάξει. Αν γίνει κάποια ερώτηση, μπορείτε να, ρωτήσετε, να απαντήσετε όχι. Λοιπόν, 39 υπέρ κατά, ποιες απορρίπτονται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 32 παρακαλώ την 32 πέρας και εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 όχι καταπίπτει Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 καταπίπτει. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε 43 παρακαλώ. Τη 43. Πέρας. Ο, ζητώ συγγνώμη, πήγα πολύ γρήγορα. 44 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, να ελέγξουμε την 5. Πέρας. Και απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47, όχι, καταπίπτει. 48 επίσης. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και 57 υπέρ όχι, όχι ζητώ συγγνώμη καταβλήτη υπάρχει μόνο 9 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να την ελέγξουμε. Την 9. Πέρα Και εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές. Ποιος είναι υπέρ της 58, ξαναλέει η πρόεδρο. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά, όχι καταπίπτει 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται να ελέγξουμε την 64 πέρας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. 65. No. Κάτι λέγεται εκτός μικροφώνου. Κοιτάξτε, το σύστημα το δείχνει αμέσως όταν έχουμε ε, πολλές ψήφους. Διεξάγεται μια συνομιλία εκτός μικροφώνου. No, they don't vote. No, no, no. Mr. Novakov is not voting. Ο κύριος Νοβάκοφ δεν, δεν ψηφίζει. Η κυρία Λικοπέτση ούτε. η κυρία Πιτέρα ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Όχι, όχι, λέει η Πρόεδρος, σε κάτι που δεν ακούμε. Η κυρία Σμιτ, Σαλαφράγκα, Ματριτσέλο, Ντόιτς, Ρουλ Μάγια, 8. Ψηφίζουμε. No, don't, don't worry. Don't, no, no, don't. 65 in favor. Συνεχίζει η πρόεδρος. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε την 66. The check is over. Πέρασε. Εγκρίνεται.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 Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 80. Μάλλον απορρίπτεται. Όχι, όχι, όχι. Σαφώς απορρίπτεται. Δεν έχουμε έλεγχο, λέει τώρα η πρόεδρος. 21 υπέρ κατά εγκρίνεται, 22 υπέρ κατά εγκρίνεται, 81 καταπίπτει, 23 υπέρ κατά εγκρίνεται, 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφοφορία για το σύνολο της νομοδότησης άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 18-2 συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, παρακαλώ να το κάνουν το συντομότερο δυνατό και όσο πιο σιωπηρά μπορούν, για να συνεχίσουμε. Η κυρία Γλίκο Γκάιτφελς, ως ε, υποψήφια της Ουγγαρίας για, την, ε, για τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, Πολύ χαιρόμαστε που επιτέλους ονομάστηκε υποψήφιος στην Ουγγαρία. Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφε. Καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Τη διαδικασία τη γνωρίζετε, όπως πάντα. Η υποψήφια, ε, στην προκειμένη περίπτωση, μας συστήνεται Συνάδελφο Τάραντιν, ο θα λάβει μετά το λόγο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εφόσον το επιθυμούν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Πρόεδρε, κύριε Τάραντ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερη τιμή που μπορώ να είμαι ενώπιον τη Επιτροπή σα σήμερα για να σα παρουσιάσω και να υποστηρίξω την υποψηφιότητά μου για μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ουσιαστικά το θέμα είναι οι δεξιότητε, οι ικανότητε και η εκπλήρωση των απαιτήσεων τη θέση, ε, η ανεξαρτησία, η λήψη συγκρού συμφερόντων. Θα ήθελα λοιπόν εν συντομία να σα παρουσιάσω το υπόβαθρο, το επαγγελματικό, την εμπειρία μου και τα σχέδιά μου για το μέλλον σε σχέση με τη θέση αυτή. Στην επαγγελματική μου ζωή πάντοτε προσπαθούσα να εμβαθύνω τις γνώσεις μου και να αποκτήσω περαιτέρω δεξιότητες ως πιστοποιημένη ηλέκτρια, φοροτεχνικός και σύμβουλος σε ευρωπαϊκό επίπεδο Σταμάτησα τις καθημερινές μου δραστηριότητε όταν ε, έγινα ευρωβουλευτής. Συνέχισα όμως το επαγγελματικό μου έργο ως μέλος των Επιτροπών Ήμικο και ΕΚΟΝ. Επίσης ήμουν υπεύθυνη για το πάνελ λογιστικού ελέγχου και την πρόσβαση στα έγγραφα ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Το Δεκέμβριο του 2016 τη habilitation degree σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του δυναμικού τη νέα αγορά. Αυτά μέχρι ε, τώρα τι έχω κάνει και τώρα θα σας πω τι θα κάνω αν γίνω μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι η φυστάμενη έλεγχη γίνονται με σωστό τρόπο, εφαρμόζονται σωστά και αυτό είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της συνολικά. με τις εκθέσεις του ελεγκτικό συνέδριο, ε, ελέγχει τα κρατημέλη, βλέπει τι αδυναμίες υπάρχουν, ε, τι έλεγχοι πρέπει να γίνουν. Και με τις γνωμοδοτήσεις του κατευθύνει και τους ευρωβουλευτές ε, και δημιουργεί ευαισθητοποίηση για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Και με τις μελέτες, με τις αναλύσεις που μπορεί να διαβάσει κανείς στο διαδίκτυο, μπορεί να διαφωτιστεί για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνετε για να σας αναφέρω κάποιες σκέψεις και να σας μιλήσω κάποιες τεχνικές επιχειρησιακές ε, εξελίξεις με βάση την εμπειρία που είχα ως ε, ελεγκτρία πριν γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω μάλιστα καταρτήσει πολλές ε, δημοσιονομικές γνωμοδοτήσεις ε, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πιο σαφή, πιο ακριβή μεθοδολογία, γιατί αυτό θα διευκολύνει το έργο των ευρωβουλευτών, θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα τις δημοσιονομικές διαδικασίες και τη σύνθεση, τη του προπολογισμού. Υπάρχει συνδιαχείριση ήδη πληροφορίες των κρατών μελών θα καθορίσουν και την ποιότητα των αξιολογήσεων. Επομένως, τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι έτοιμα να δίνουν σαφείς επίκαιρες επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες και θα πρέπει να παρακολουθεί και το ελεγκτικό συνέδριο της εκτέλεση των συστάσεων που έχει κάνει σε αιτήσιες εκθέσεις απαλλαγήση. Η αυτόματη συγκέντρωση είναι κάτι θετικό στι ειδικέ εκθέσει για να μπορέσει να τι αξιοποιήσει καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτέ πολύτιμε εκθέσει πολύ συχνά δεν παίρνουν την προσοχή που του αξίζει. Επίση, θεωρώ ότι η νομοδοτοήσεις του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά και τη, δουλειά που κάνουμε εδώ είναι κάτι πολύ αναγκαίο και χρήσιμο. Πλήρη λογοδοσία. Συμμόρφωση με τους κανόνες για τα χρηματοδοτόμενα από την Ένωση project. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα κανόνων και ότι είναι οι πιο ενδεδειγμένοι κανόνες. Πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε καλύτερα τη σχέση του ωφέλους και να έχουμε ελέγχους απόδοσης, γιατί αυτό θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Επίσης, είμαι πεπισμένη ότι στοχευμένη διαχείριση της έρευνας απαιτεί και αυτή ειδική προσοχή. Ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε κατά πόσο η προσθέμενη αξία των ευρωπαϊκών κονδύλων έχει ληφθεί υπόψη στη φάση του σχεδιασμού. Στο πλαίσιο του ποιητικού ελέγχου τώρα, θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά όλα τα μέτρα που είναι αποτέλεσμα των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα, μπορεί, θα πρέπει το συνέδριο να μπορεί να βασίζεται στις εθνικές εποπτικές αρχές για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις και αχρία στο γραφειοκρατικό ή διοικητικό άχθος. Υπάρχει μια μακρά παράδοση συνεργασίας στο πλαίσιο του Ιντεσάι. Έχουν υπάρξει σημαντικέ βελτιώσεις στο τομέα τη τυποποίηση. Επίσης, είναι σημαντικό τα αποτελέσματα των εθνικών ελέγχων να ε, ενσωματώνονται στι δραστηριότητε του ελεγκτικού συνεδρίου. Ταυτόχρονα υπάρχουν ευκαιρίε και για δραστηριότητε κοινού ελέγχου. Κατά την άποψή μου, μια άλλη σημαντική προτεραιότητα θα είναι οι εθνικέ αρχέ ελέγχου να εστιάσουν περισσότερο στον έλεγχο τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Πολύ καλό παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών είναι η συζήτηση των εκθέσεων αυτών στα εθνικά κοινοβούλια και η διατύπωση συμπερασμάτων. Κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων στο μέλλον. Ευρύτερη διάδοση λοιπόν των πιστοποιητικών ελέγχων θα μπορούσε να είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι το Ελεκτικό Συνέδριο είναι ένας στενός σύμμαχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε την ίδια αποστολή, δηλαδή την διαφύλαξη των συμφερόντων των φορολογμένων και των πολιτών της Ένωσης. Σε περίπτωση που ε, οριστώ ανεξάρτητο, αμερόληπτο μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια στα αναλυτικά, εποπτικά μου και λογιστικά μου καθήκοντα για να υπηρετήσω τις ανάγκες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διευκολύνω την ομαλή χρήση των πόρων της Ένωσης και να προωθήσω τη βιωσιμότητα της χρηστής διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω και στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή. Ο εισηγητή, ε, Τάραντ, έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο έκθεσης με βάση το ερωτηματολόγιο το οποίο σας είχαμε αποστείλει. Έχει το λόγο. Κύριε Τάραντ, παρακαλώ. Ε, sorry, Madam President, I sort of was cut off from Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την υποψήφια για το ελληνικό συνεδρίο και να πω ότι παρότι η ζωή είναι πολύ ήρεμη και μέχρι και βαρετή στο Λουξεμβούργο, μπορείτε να βρείτε μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θέλω να προσβάλλω το Λουξεμβούργο. Είναι μικρή χώρα, αλλά μικρή σε σχέση με την Ουγγαρία απλώς. Έχω μια-δυο ερωτήσεις πάντοτε για τους υποψηφίους. Με εσά θέλω να ξεκινήσω με μια ιδιαίτερη ερώτηση ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πόσο σκληροί και αυστηροί θα είστε προς τις ε, διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δαπανών στο Κοινοβούλιο. Επί τη σας εδώ. Η δεύτερη ερώτηση είναι πιο φιλοσοφική. Κατά την άποψή μου δεν απαγορεύεται να κάνει κανείς μια διαφορετική δουλειά μετά την πολιτική του θητεία, αλλά αυτό μας ξαναφέρνει στο Κοινοβούλιο. Όταν θα ελέγχετε τις δραστηριότητες μας, πώς θα μπορέσετε να διακρίνετε μεταξύ των δύο ρόλων σας. Και τρίτον, και πιο σημαντικό, ίσως να μην καταλήξει αυτό το θέμα στο γραφείο σας στο Λουξεμβούργο Αλλά από πού θα, μετα... θα μετακομίσει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο από τη Βουδαπέστη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσής του ε, και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις συνομιλίες που είχαμε ήδη. Η πρώτη σας ερώτηση είχε να κάνει με το πώς θα συνεχίσω τη σταδιοδρομία μου ανεξάρτητη ε, μετά τη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως σας είπα και εισαγωγικά, ήμουν αντιπρόεδρος ε, του, της Ελεγκτικής Επιτροπής Δηλαδή έχω ασχοληθεί και με τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί χρειάστηκε ανεξαρτησία και αμεροληψία και νομίζω ότι σχετικά καλά τα πήγαμε. Και νομίζω ότι δεν χωρά καμιά αμφιβολία ε, ως προς την ανεξαρτησία και την αμεροληψία μου. Ούτε πολιτικές ήταν οι αποφάσεις, ούτε μονομερείς. Υπάρχει ένα θέμα που με απασχόλησε ήδη και αυτό είναι ο προπολογισμό του 2017 που μπορεί να είναι ακαθόδης και λεπτό. Διότι από κοινού όλοι μαζί στο Κοινοβούλιο αποφασίσαμε τον προπολογισμό του 2017, το ψηφίσαμε και ως μέλος του Προεδρείου ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχα στη λήψη των αποφάσεων αυτών. Και νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό ε, να ε, ελέγξω την εκτέλεση του προπολογισμού του 2017. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί δεν θα ανήκω ε, στο συγκεκριμένο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου που ασχολείται με τον έλεγχο αυτό. Μέχρι τώρα πάντως φρόντιζα ανέκαθεν να παραμένω ανεξάρτητη και αντικειμενική σε όλα τα θέματα. Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με την πρόσβαση στα έγγραφα, Φέρυπιν. Ανέκαθεν εφρόντιζα όταν κάνουν κάποιες ερωτήσεις ε, Ούγγροι πολίτες να μην είμαι εγώ εκείνη που θα λάβει την ε, σχετική απόφαση. Και πάντα φρόντιζα να παραμείνω ανεξάρτητη και το ανέθετα σε κάποιον άλλον. Σε ό,τι αφορά ε, το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης, ελπίζω να παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα στη Βουδαπέστη και να λειτουργεί και το λέω και ως πανεπιστημιακή αυτό και ως πανεπιστημιακή διδάσκαλα. Ο εισηγητής έχει συμπληρωματικές ερωτήσεις. Uh, no, you, Όχι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα μέλη λοιπόν, η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ σχετικά με την υποψήφια, καθότι είχατε χρηματίσει και ελέγκτρια και φοροτεχνικός, ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν συμμετείχατε ποτέ στην Επιτροπή μας παρότι πράγματι ο συνάδελφός σας ο κύριος Ντοίτς είναι πολύ ενεργός εδώ αλλά πέραν αυτού θα γνωρίζετε ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο για το ελεγκτικό συνέδριο αλλά συνολικά για την Ένωση είναι η προσπάθεια θέσπισης προϋπολογισμού επί τη βάση των αποτελεσμάτων το οποίο σημαίνει ότι ο έλεγχος όχι μόνο του ελεκτικού συνεδρίου, των λογαριασμών, των ισολογισμών και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού πρέπει να εμβαθύνει στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. Και πρέπει να πω ότι με ανησυχεί ότι το κόμμα σας και η κυβέρνηση του κόμματός σας στη χώρα σας επιδεικνύει έναν αντιευρωπαϊσμό αλλά κυρίως μια αντίθεση προς πολιτικές ε, τόσο σημαντικές Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εκείνη της ένταξης των μεταναστών και της ε, ενσωμάτωσης ή της υποδοχής καλύτερα των προσφύγων. Εκτός λοιπόν από την ανεξαρτησία σας, μας χρειάζονται και τέτοιου είδους ε, ενδείξεις, πτυχές ώστε να εξασφαλίσουμε όχι μόνο ότι θα εκτελούμε σωστά τον προϋπολογισμό, αλλά το ελεγκτικό συνάδριο πολύ συχνά κάποιες φορές μας λέει ότι καλώς δαπανίσατε ή όχι, άλλες φορές μας λέει ότι τα χ ή ψ κονδύλια για την τάδε πολιτική είναι ή δεν είναι αρκετά και η γνώμη σας πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητη από την ε, ενεργό πολιτική σας ζωή που είναι που έχετε επιδείξει μια έντονη πολιτική δραστηριότητα και είναι φυσιολογικό αυτό βεβαίω. Επίσης, τι άποψη έχετε, θα ήθελα να ξέρω, για την ανάμεξη μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων συνοχής με τα κονδύλια του ΕΦΣΙ του σχεδίου Juncker. Είναι ένα θέμα που συζητείτε πολύ αυτή τη στιγμή. Ήθελα να καταλάβω αν έχετε μια τοποθέτηση από αυτό. Και Τέλος, καθότι πολύ καλά είπε η Πρόεδρος, ένα χρόνο τώρα περιμένουμε το διορισμό του ογκρικού μέλους και πολύ μας ικανοποιεί το γεγονός ότι είστε εσείς, είστε γυναίκα, είστε συνάδελφος, σας γνωρίζουμε. Θα είναι από 1η Μαΐου ή από 1η Ιουνίου που θα ενταχθείτε στην υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα Σέντερ για τις ερωτήσεις σας αυτές. Για να είμαι πολύ τους ειλικρινής, δεν ήμουν εγώ η πρώτη υποψήφια, ε, αλλά η τελευταία, δηλαδή το όνομά μου επικράτησε τελικά χωρίς να είμαι η πρώτη επιλογή της Ουγγαρίας για το ελεγκτικό συνέδριο. Παρ' όλα αυτά χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, η ε, δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά με ικανοποίησε πάρα πολύ. Είχαμε ένα στόχο να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις και σε υψηλά πόστα. Και ε, μετά την ε, επιτυχημένη, ελπίζω, ακρόαση, έχω την ελπίδα να ε, διοριστεί ακόμα μια γυναίκα στο ελεγκτικό συνέδριο. Βέβαια, απέχουμε ακόμα πόρο από την ισότητα των φύλων σε ό,τι αφορά τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Για το δεύτερο που με ρωτήσατε, που μπορώ να δραστηριοποιηθώ, αυτό θα εξαρτηθεί από το Συμβούλιο. Και φυσικά θα σεβαστώ την απόφαση του Συμβουλίου και θα προχωρήσω ανάλογα. Εγώ με μεγάλη χαρά ε, θα ήμουν μέλος ε, της Επιτροπής σας Ελέγχου του προπολογισμού ως ε, φοροτεχνικός και λογίστρια. Αλλά ο κύριος Τόμας Ντόιτς ήταν βουλευτής πριν από μένα και μέλος στην Επιτροπή σας και δεν ήταν κομψό να τον εκτοπίσω. Και επίσης ενδιαφερόμουν και για άλλες επιτροπές. Ε, για την Οικονομική ε, και Νομισματική Επιτροπή, όπου δεν υπήρχε ο Ούγγρος βουλευτής τότε και αντιστοιχούσε και στη δική μου επαγγελματική δραστηριότητα, ακόμα και στην Επιτροπή Νέας Αγοράς, στην ΙΜΚΟ, ε, που γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα και με ενδιέφερε πάρα πολύ και είναι και ένα τεράστιο δυναμικό αυτό που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί πλήρως, ούτε εξαντληθεί. Γιατί χρειάζεται να γίνουν περισσότερα βήματα και να ληφθούν και άλλα μέτρα. Για την δεύτερη ερώτησή σας τώρα, πώς θα έχουμε αποτέλεσμα eh, στις εργασίες μας. Κοιτάξτε, δεν αρκεί να κάνουμε σε τακτά ε, χρονικά διαστήματα ελέγχους κατά πόσο τηρούνται και εκτελούνται όλα σωστά και δεν παραβιάζεται η νομοθεσία. Αυτό είναι το λιγότερο. Ε, το μεγάλο ερώτημα είναι ε, αν θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Γιατί μέχρι σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα υπολείπονται των στόχων. Για το 2020 έχουμε ωραίους στόχους και ε, μεγαλεπίβολους, τους οποίους δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να υλοποιήσουμε. Γι' αυτό ε, τι πρεσβεύω ότι θα πρέπει συνέχεια όλο και περισσότερο να γίνονται λογιστικοί έλεγχοι των επιδόσεων. Ε, Βεβαίω θα ελέγχουμε και το σύνομο, αν υπάρχουν παρατυπίες ή όχι. Αλλά ε, χρειαζόμαστε καλούς δείχτες για να μετράμε τις επιδόσεις. Αν θυμάστε κάποιες περιπτώσεις ε, που εγκρίναμε τέτοιες εκθέσεις, το πρόβλημα ποιο ήταν τότε. Ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούσαν πάρα πολλούς δείκτες, ποσοτικούς και ποιοτικούς μπορούμε να την αναλύσουμε έτσι την επίδοση και έτσι δηλαδή. Αλλά αν δεν έχουμε καλούς δείκτες αξιόπιστους δεν μπορούμε να ε, ε, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλές συγκρίσεις από χώρα σε χώρα ή από τη μια χρονική στιγμή στην άλλη. Αυτούς τους ελέγχους θέλουμε να κάνουμε λοιπόν των επιδόσεων και όχι μόνο των, τους τυπικούς. Αυτό που μας νοιάζει είναι κάθε φορά που επενδύουμε ή δαπανούμε ένα ευρώ, ποια είναι η απόδοση, πόσο τόπο πιάνει και τι μας αποφέρει. Ξέρω ότι η τελευταία έκθεση της, ε, του ελεκτικού συνεδρίου, μάλλον που αναφέρατε κι εσείς, για τις συμφωνίες εταιρικών σχέσεων, διαπιστώνει προβλήματα. Χρειάζεται βελτίωση και εναρμόνιση και των δικτών και όλης της ορολογίας. Διότι έχει διαφορά. Πραγματικά τους ίδιους όρους τους χρησιμοποιούν διαφορετικά και τους ερμηνεύουν διαφορετικά τα κράτη-μέλη για την ανεξαρτησία. Δεν τίθεται καν αυτό το θέμα ε, να μεροληπτήσω. Καθ' όλη τη διάρκεια, μάλλον πριν την πολιτική μου στραδιοδρομία, ε, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο. Είχα βέβαια την προσωπική μου ε, γνώμη, αλλά ο Δής ποτέ αμφισβήτησε την ανεξαρτησία μου και την αντικειμενικότητά μου. Ούτε ήξεραν οι φοιτητέ ε, τις πολιτικές μου πεπιθήσεις, ούτε ήθελαν να τους τις επιβάλλω. Επάγγελμα ήταν. Και το ελεκτικό συνέδριο είναι ε, μια θέση όπου εργάζονται επαγγελματίες με ανεξαρτησία και μεροληψία. Επίσης όταν διατέλεσα ε, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποτέ δεν θα ε, είδατε από μένα υπερβολές ή πολιτικές έτσι, οξύσεις. Δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων. Σε περίπτωση που είναι θετική η έκβαση της σημερινής ακρόασης και η δική σας γνωμοδότηση γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσα να λάβω αυτή τη θέση. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Βεβαίω εσείς δεν έχετε παρακολουθήσει τη σταδιοδρομία μου, αλλά μπορεί να διαπιστώσετε ότι από τον επίσημο διορισμό μου ως υποψήφια δεν έχω προβεί σε καμία δήλωση που θα μπορούσε να ε, πλήξει την ανεξαρτησία μου. Ελπίζω να απάντησα σε όλε τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα 8 συναδέλφου στον κατάλογο των ομιλητών. Ε, εντάξει, παρακαλώ να είστε σύντομοι όσο γίνεται και υποψήφια. Ο συνάδελφο Νόβακοφ. Thank you, Chair. I'll be brief. I'm always positive when colleague Είναι θετικό να ορίζεται ένα συνάδελφος, ευρωβουλευτής, ε ως υποψήφιος ε, για το ελεγκτικό συνέδριο. Κατά την άποψή μου τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι είναι αυτό ένα ασφαλή τρόπο να βελτιώσουμε τι σχέσει μεταξύ ελεγκτικού συνεδρίου και κοινοβουλίου και νομίζω πω υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Τώρα, για τι ερωτήσει και τα σχόλια που ακολουθούν, ε, εκπροσωπώ και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Σαρβαμά, και, το, ε, και εκφραζώ και τις προσωπικές μου απόψει. Και ο κύριο Σαρβαμά δεν μπορούσε να είναι εδώ στο βιογραφικό σας λοιπόν και στις γραπτές σας απαντήσεις, ε, κύριε Γκάλ Πέλτς, ε, αλλά και με το αξιώμα της Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου και ως βουλευτής, δείξατε ότι έχετε τεταμένη γνώση του χρηματοψηφιακού συστήματος και των ελεκτικών διαδικασιών. Παρομοίως δείξατε ότι είστε ικανοί να μπορέσετε να αναπτύξετε τα στήματα αυτά ε, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και επιλέγοντας τις πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Ε, θα ήθελα ωστόσο να σας ε, ζητήσω να μου πείτε πώς θα βελτιώσετε συγκεκριμένα τις διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο το ελεγκτικό συνέδριο εκτελεί τα καθήκοντά του σε περίπτωση που επιλέγετε για τη θέση αυτή. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία απαλλαγή και άλλες μεθόδους παρακολούθησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα πρέπει ε, να λαμβάνουμε ποιοτικέ πληροφορίε για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων τη Ένωση, ώστε να μπορούμε να αναπτύσσουμε πολιτικέ και κανόνε ε, για το πώ δαπανώνται τα κονδύλια τη Ένωση. Ποιε συγκεκριμένε εξελίξει ε, θα δρομολογούσατε με βάση την, τον έλεγχο βάση επιδόσεων. Δεύτερον, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια ο αριθμός ε, των εκθέσεων. Το 2007 ήταν 9 μόνο και φέτος είναι 36, στον πέρυσι 36. Ποιο είναι ο βέλτιστος αριθμός ε, των εκθέσεων, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί και να μην μπορεί καν να επεξεργαστεί ετησίω όλα αυτέ τι εκθέσει, γιατί η ποιότητα νομίζουμε ότι πρέπει να είναι πιο καθοριστικό παράγοντα από την ποσότητα. Αν συμφωνείτε, τι βελτιώσει θα προβλέπατε. Τέλος, η Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού του Κοινοβουλίου δίνει μεγάλη έμφαση στη στενή σχέση μεταξύ των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου. Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και διασύνδεση, διασυνδέσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς θα εκμεταλλευτείτε το πλεονέκτημα αυτό για να βελτιώσετε ακόμη περισσότερο τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πέλτς, ε, ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Νόβακοφ για αυτές τις ερωτήσεις. Και βέβαια και τον κύριο Σαρβαμά θέλω να ευχαριστήσω αφού από κοινού ε, έχετε διατυπώσει αυτές τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με την πρώτη ερώτηση σε ό,τι αφορά ε, την, τον έλεγχο της αποδοτικότητας και τον έλεγχο βάση επιδόσεων. Νομίζω ότι έχει ληφθεί μια πολύ καλή απόφαση από το ελεγκτικό συνέδριο όταν διαπίστωσε ότι θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτόν τον έλεγχο ε, της αποτελεσματικότητας. Ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο λοιπόν και την παρακολούθηση των επιδόσεων, σίγουρα χρειάζονται ποιοτικέ πληροφορίες που πρέπει να διαθέσουν τα κράτη-μέλη. Βέβαια, αυτό είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Θα πρέπει να δίνουν ε, τις επίκαιρες ε, και ενδεδειγμένες πληροφορίες εγκαίρως στα κράτη-μέλη και όσο το δυνατόν ε, πιο γρήγορα θα πρέπει οι ελεκτές να έχουν λάβει αυτές τις πληροφορίες ώστε να μπορούν να φέρουν σε πέρα αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαν να, να ε, φέρουν σε πέρα σωστά τις εργασίες τους οι ελεγκτές και να πρόκειται σωστά συμπεράσματα. Από την έννοια αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, νομίζω κάνει και ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. με το ολοκληρωμένο πακέτο ελέγχου και νομίζω ότι οι έλεγχοι επιδόσεων και τα λοιπά θα βελτιωθούν και στο μέλλον. Θα με βελτιώνονται όλο και περισσότερο. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω το εξή Έλεγχοι επιδόσεων και τα λοιπά ποτέ δεν θα πρέπει να ε, έρχονται σε βάρος ε, του έλεγχου συμμόρφωσης. Πριν από λίγο μίλησα ε, για τους ε, κινδύνους ό,τι αφορά το συντελεστή σφάλματος. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται σίγουρα να υπάρχει όμως. Μόνο να τα κάνουν τον έχω από αυτή την πλευρά. Δεν είναι καλό χρόνο το χρόνο να ανακαλύπτουμε νέες μεθόδους με τις οποίες θα φέρουμε σε πέρας ε, τους ελέγχους, διότι δεν θα έχουμε παρκή χρόνο για να κάνω σωστά ε, τους ελέγχους. Επίσης είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να επισέλθουμε σε μεγάλες λεπτομέρειες. Χρειαζόμαστε δείκτες με τους οποίους θα μπορούμε να συλλέγουμε σχετικά εύκολα τις πληροφορίες. Και θα πρέπει να πρόκειται για πληροφορίες που εύκολα μπορεί κανείς να τις ε, εντοπίσει μέσα στο σύστημα και σε ό,τι αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και στον έλεγχο ε, υπάρχει κάτι το οποίο έλειπε, αν θέλετε, ένα στοιχείο σε σχέση με το feedback, α, τον έλεγχο, δηλαδή από το κοινοβούλιο προς το, από το ε, ε συνέδριο προς το κοινοβούλιο και το αντίστροφο. Είναι πάρα πολύ σημαντική σχέση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Γνωρίζουν πολύ καλά οι ευρωβουλευτές πόσο σημαντικό είναι το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου. Επίσης, εξίσου ε, σημαντικό είναι το έργο του Κοινοβουλίου για το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου. Χρειάζεται λοιπόν αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Και θα έλεγα ότι ίσως και καθημερινή επαφή ε, δεν θα έβλαπτε. Τώρα, είδα τις ειδικές εκθέσεις ε, και πόσο έχει πραγματικά αυξηθεί ο αριθμός αυτών των ειδικών εκθέσεων. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Φυσικά δεν θα ήθελα ε, να ξεκινήσω ασκώντας κριτική αμέσως στο Ελληνικό Συνδρίο μόλις αναλάβω καθήκοντα. Ίσως καλό θα ήταν υπάρχει θεματική ε, ομαδοποίηση των ειδικών εκθέσεων. Έχουμε 36 τις οποίες τέσσερις έχουν να κάνουν παραδείγματος με την ανεργία, που είναι ένα σημαντικό θέμα βέβαια, ιδίω σε σχέση με την ανεργία των νέων. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε δημιουργήσει την εγγύηση για την νεολαία και υπάρχει και ένα σημαντικό ποσό που προβλέπεται στον ε, προϋπολογισμό 6,4 δις για το θέμα αυτό. Άρα, σίγουρα το μέα τη ανεργία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια άνεργοι στην, ε, ε, νέοι στην Ευρώπη που δεν μπορούν να, να βρουν θέση εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν νομίζω όμω ότι θα βοηθήσει την κατάσταση να βελτιωθεί η σύνταξη πολύ περισσότερων ειδικών εκθέσεων για το θέμα αυτό. Ίσως καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρξει μια θεματική συγκέντρωση των ειδικών εκθέσεων. Και ένα άλλο θέμα είναι το χρονοδιάγραμμα. Ε, θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη, το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι ειδικέ εκθέσει όταν αυτέ είναι επίκαιρε. Δεν χάνουν δηλαδή το στοιχείο τη επικαιρότητα. Μπορούμε να το δούμε αυτό βέβαια τις μεθόδους, το χρονοδιάγραμμα για τη ε, τις για τη σύνταξη μιας ειδικής έκθεσης. Παραδείγματος χάρη, ειδική έκθεση για τα προβλήματα της μετανάστευσης. Όταν ήρθε αυτή η ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, δεν, δεν ήταν πια επίκαιρη. Ε, είχαν αλλάξει τα νούμερα, δεν ήταν πια επίκαιρα και το καθεξής. Άρα θα πρέπει να είναι επίκαιρο κατά το δυνατόν πληροφορίε ε, και το περιεχόμενο των δικών θέσεων. Αυτό κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου, για να λειτουργεί σωστά αυτή η συνεργασία, μάλλον αν λειτουργεί καλά η συνεργασία, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και τα διαθεσμικά όργανα και θα μπορούμε επίση να φέρουμε σε πέρα καλύτερα και τα καθήκοντά μα και να εγγυηθούμε την ε, τη σωστή ε, οικονομική διαχείριση. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ευθύ εξ αρχή ότι ένα θετικό στοιχείο είναι ότι έχουμε μια γυναίκα υποψήφιο. Δεν είχαμε αρκε... αρκετές. Και με το άνω του μισού του πληθυσμού που είναι γυναίκες αναρωτιέται κανείς γιατί δεν βλέπουμε περισσότερες υποψήφιες και μέλη γενικώ Τώρα, είσαστε μέλος του κόμματος Φιντές, δεν το προφέρω σωστά. Ήσασταν και αντιπρόεδρος του κόμματος αυτού για τέσσερα χρόνια μέχρι το 2010. Και θα ανησυχούσε ιδιαίτερα να υπερψηφίσω οποιοδήποτε μέλος του κόμματος εκείνου δεδομένων κάποιων δηλώσεων που έχουμε ακούσει από τον ηγέτη σας, όπως οποιαδήποτε πολιτική μετανάστευση είναι απειλή για την ασφάλεια και ότι η μετανάστευση είναι δηλητήριο και δεν πρέπει να το καταπιούμε το δηλητήριο αυτό. Αυτά λέει ο ηγέτης Με αυτά συμφωνείτε και αν δεν συμφωνείτε, τι έχετε κάνει για να τα αντικρούσετε. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια και ιδιαίτερα ε, στην οικογένεια της γυναίκας μου, 19 εκ των 20 που χρειάστηκε να πάνε στο Λονδίνο για οικονομικούς λόγους, ε, φαντάζομαι ότι βάσει της ιδεολογίας σας είμαστε οι χειρότεροι, οικονομικοί μετανάστες. Και τι θα έπρεπε να γίνει με την αδελφή της γυναίκας μου που έχει γεννηθεί στο Λονδίνο αλλά εσείς ονομάζετε ανθρώπους σαν την αδερφή της γυναίκας μου δηλητήριο, απειλή για την ασφάλεια. Γιατί θα έπρεπε να σας υπερψηφίσω. Παρατήρησα ότι συμπεριφερθήκατε με κάποια συμπόνια με τον συνάδελφό σας και δεν θέλατε να τον διώξετε από τη θέση του αλλά θέλετε να διώξετε τους μετανάστες ακόμα και αν δεν έχουν αρκετό φαγητό. Κύριε Πρόεδρος, θα ήθελα να θυμίσω ότι συζητάμε με την κυρία Γκάλ Πέλτς και αυτό είναι το θέμα και όχι ο Ούγγρος Πρωθυπουργός. Και για μένα έχει σημασία να παραμείνουμε στο θέμα μας. Η κυρία Γκάλ Πέλτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κύριε Φλάναγκαν για τα όσα είπατε. Έχω πολύ την κατανόηση για τα λεγόμενά σας. Και βεβαίως χαίρομαι που μπορώ να σας απαντήσω ως γυναίκα για τα θέματα της ε, ίσης εκπροσώπησης. Για να διατηρηθεί και η ισορροπία έχω φορέσει παντελόνι σήμερα, έτσι, για να ε, χαριτολογήσω. αντιπρόεδρος του ΦΙΝΤΕΣ είμαι από το 2005, όχι τα τελευταία χρόνια. Είμαι αντιπρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος ε, του τμήματος γυναικών. Και μπορώ να σας πω πόσα έχω επιτύχει ε, και στην οικογενειακή πολιτική και άλλα που είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε από τις γραπτές μου απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Και έχω κάθε λόγο να είμαι υπερήφανη για όλα αυτά τα επιτεύγματά μου. Φυσικά δεν ταυτίζονται οι απόψει όλων για όλα τα θέματα. Αυτό που έχει σημασία σήμερα στην παρούσα ακρόαση για μένα είναι ε, να μοιραστώ μαζί σας ότι έχουμε συναντήληψη για τα θέματα αυτά, τα αντικειμενικά, τα οικονομικά και του ελεκτικού συνεδρίου. Πολιτικά μπορεί να μην συμφωνούμε, που δεν συμφωνούμε κιόλα. αλλά αυτό θα ήταν άστοχο ε, να το συζητούμε τώρα για το ελεγκτικό συνέδριο. Και νομίζω ότι από τη δουλειά μου μέχρι τώρα έχω αποδείξει ε, και μπορείτε να το θεωρείτε ως εγγύηση ποια είναι η στάση μου παραμένω ανεξάρτητη, ικανή, αμερόληπτη, χωρίς την παραμικρή επιρροή θα ασκήσω τα καθήκοντά μου στο μέλλον όπως έκανα και στο παρελθόν. Και μπορώ να δεχτώ επίσης να με καταψηφίσετε. Αλλά παρακαλώ ε, να σκεφτούμε περί τίνος πρόκειται στην παρούσα ακρόαση. Είναι ένα θέμα ε, ειδικό αντικειμενικό τεχνικό δεν έχω τίποτα στη σταδιοδρομία μου που να μπορεί κανείς να μου προσάψει και παρακαλώ να με εμπιστευτείτε. Με την ίδια αντικειμενικότητα ε, θα συνεχίσω τη δουλειά μου. Περί αυτού πρόκειται. Για το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν είναι θέμα μετανάστευσης. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μία από τις τέσσερις βασικές κυκλοφορίες ε, ελευθερία, συγγνώμη. Το ποιο θα μεταβεί από τη μία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια άλλη για να αναζητήσει δουλειά δεν είναι πρόβλημα. Αν ήταν στο χέρι μου να το αποφασίσω εγώ, θα παρότρινα τους νέους να ε, ε πάνε σε ένα άλλο κράτος μέλος για να βρουν δουλειά, γιατί αυτό είναι προς όφελος όλων των κρατών μελών. Αν δείτε τα ποσοστά ελεύθερη κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συγκρίνεται με τις Ηνωμένε Πολιτείε. δεν είναι καθόλου υψηλό το ποσοστό αυτό στην Ευρώπη. Το αντίθετο μάλιστα. Έχουμε νέους ανέργους, οι οποίοι πολύ καλά θα έκαναν να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό. 46 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Ε, όσα χρήματα και να δώσουμε στους νέους δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν. Αλλά δεν μπορεί να αποφυτούν από το σχολείο και να μην βρίσκουν δουλειά και να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βρουν δουλειά. Φυσικά θα πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την ελευθερία της κυκλοφορίας και των νέων μας. Πάντως αντικειμενική στη δουλειά μου θα είμαι και μπορώ να σα το διαβεβαιώσω. να Σαναβουστάς από του πρασίνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ την υποψήφια, όπως και ο κύριος Φλάναγκαν. Χαίρομαι πάρα πολύ που η εγκρική κυβέρνηση πρότεινε γυναίκα, γιατί πραγματικά μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει και στο ελεκτικό συνέδριο σε εκπροσώπηση. Κυρία μου, είστε μέλος του ΦΙΝΤΕΣ, ε, το κόμμα της πλειοψηφίας και της κυβέρνησης στην Ουγγαρία, η οποία δεν διακρίνεται σήμερα ε, από την αγάπη της προς τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Λέτε ότι η σημερινή ακρόαση έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένα θέματα, το ξέρω, αλλά η κυβέρνησή σας δηλώνει ότι η στήριξη των ΜΚΟ από το εξωτερικό μπορεί να απειλεί την εσωτερική ασφάλεια της Ουγγαρίας. Εγώ διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί. Οικονομικά ε, δηλαδή έχουμε ροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα προς μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Και σας ερωτώ, συμφωνείτε εσείς με τις δηλώσεις ε, της πλειοψηφίας της χώρας σας της κυβέρνησης ότι η οικονομική στήριξη από το εξωτερικό προς μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορεί να συνιστά απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της Ουγγαρίας. Επίσης, συμφωνείτε με την άποψη που λέει όταν δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεση στήριξη σε ουγγρικές ΜΚΟ που ε, προστατεύουν τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι μπορεί αυτό να συνιστά λοιπόν απειλή για την ασφάλεια της χώρας. Αυτό που ρωτάω είναι κάτι αντικειμενικό και θα μπορούσατε ε, να μου απαντήσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στάς για την ερώτηση. Είναι πολύ βασικό το ερώτημα. Έχω να πω ότι η διαφάνεια ε, και ο επαγγελματισμό ε, σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό να είναι εγγυημένα και κατοχυρωμένα και οι ΜΚΟ διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, έχουν σημαντικά καθήκοντα και στην πολιτική μου σταδιοδρομία. Έχω ε, ξεκινήσει να εργάζομαι ε, σε μια μη κυβερνητική οργάνωση ως πρόεδρος. Ο στόχος ήταν ε, τη στήριξη, στήριξη της ανάπτυξης στη δική μου την ιδιαίτερη πατρίδα και νομίζω ότι ε, θεώρησα ότι κάτι, αυτό θα μου προσφέρει κάτι περισσότερο από το να διδάσκω στο πανεπιστήμιο. Ε, μετά, μάλιστα, εξακολούθησα ε, την ίδια κατεύθυνση. Ήμουν στα ενία μιας οργάνωσης που προσπιζόταν τα δικαιώματα των γυναικών στην Ουγγαρία. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που βρίσκονται σε μονεκτική θέση και παιδιά και οικογένειες ολόκληρες. Ο στόχος μου προσωπικά είναι να αξιοποιήσω τις επαφές μου και τα δίκτυα, τις διασυνδέσεις που έχω για να προωθήσω τους στόχους αυτούς. Είπατε κι εσείς ο ίδιος ότι είμαι μέλος του ΦΙΝΤΕΣ. Όπως βλέπετε όμως είμαι ε, μέλος και μιας μη κυβερνητική οργάνωσης. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά των κυβερνητικών οργανώσεων και αν μπορώ θα την υποστηρίξω. Μάλλον θα ξαναασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο και αν μπορώ να κάνω κάτι ή αν χρειαστεί ε, θα πρέπει να αποχωρήσω ίσως από αυτή την κυβερνητική οργάνωση. Τώρα, ε, εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε τις ΜΚΟ, κάνουν πολύ σημαντική δουλειά, αλλά εδώ δεν μιλάμε για δραστηριότητα των ΜΚΟ, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν πηγαίνει αυτή η δραστηριότητα προς την λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι χρήσιμο το έργο των ΜΚΟ. Παραδείγματος χάρη εγώ ε, που ήθελα να ε, βοηθήσω την ε, ανάπτυξη της πατρίδα ε, ως μέλος μη κυβερνητική οργάνωση. Αν έκανα κάτι που θα έβλαπτε όμως την ιδιαίτερη πατρίδα, αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα. 100% σχεδόν νομίζω τον ΜΚΟ κάνουν αυτό που κάνουν γιατί θέλουν να προσφέρουν κάτι χρήσιμο, με προσθέμενη αξία, ό,τι αφορά τα οικονομικά. Φυσικά και δεν έχουμε ε, κανένα πρόβλημα να στηρίξουμε ε, τις ε, οικονομικά πάντα της ΜΚΟ που έρχονται από το εξωτερικό. Εντελώς δεν μπορούσα να αναφέρω σε πέρα στα καθήκοντά τους. Χρειάζεται λοιπόν οικονομική υποστήριξη και από το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ήταν κακό όμως, αυτό να γίνεται με διαφανή τρόπο, η χρηματοδότηση δηλαδή, να είναι διαφανής. Και από τη δική μας την ε, ΜΚΟ, ε, φυσικά και θα χαιρόμασταν πολύ να έχουμε υποστήριξη για να πληρώσουμε καλύτερα τους στόχους μας. Και θα έπρεπε να δείξουμε και εμείς πώς χρησιμοποιούμε τους ε, πόρους, πώς αξιοποιούμε τα κονδύλια που παίρνουμε. Άρα η διαφάνεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η προβολή για να βλέπουμε ότι πραγματικά κάνουν σωστά τη δουλειά τους ε, η ΜΚΙΟ. Ο κύριος Άρνοτ από την EFTD. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπήρξαν κάποιες επίμονες ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής ε, σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι προσπαθείτε να κινηθείτε από έναν έντονα πολιτικό ρόλο σε έναν απολιτικό ρόλο. Επίσης, ε, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά σας, θα είχατε κίνδυνο να έχετε σύγκρουση με τα όσα κάνατε προηγουμένως στο Κοινοβούλιο ή στην πολιτική σας ζωή. Επομένως, πέραν των όσων είπε ο κύριος ε, Τάρεντ, <coughs> αλλά και ο κύριος Φλάναγκεν, η φύση των καθηκόντων αυτών, του ελεγκτή δηλαδή, είναι πολύ διαφορετική. Επομένω, πέραν του να πείσετε την Επιτροπή για την ε, ικανότητά σας να είστε ανεξάρτητοι και αδέκαστοι, πόσο άνετα θα αισθανθείτε αν χρειαστεί να αντιταχθείτε σε κάτι που θα θεωρήσετε εσφαλμένο στο μέλλον. και στη θητεία σας ως μέλος του Αεροκόκκινου Βουλίου είδατε, παρατηρήσατε ποτέ κάτι μέσα στην πολιτική σας ομάδα που θεωρήσατε ότι ήταν εσφαλμένο ή στο κόμμα σας το ίδιο όπου αισθανθήκατε δηλαδή ότι αυτό είναι λάθος ώστε να το εκφράσετε ανεξαρτήτως πολιτικής γραμμής της σας. Πότε πότε στο παρελθόν δηλαδή δείξατε την ικανότητά σας να εκδηλώνετε την αντίρρησή σας με κάτι που θεωρούσατε σφαλμένο. Και σε σχέση με τη μετακίνηση αυτή από τον πολιτικό βίο στο βίο του ελεγκτή, πώς θεωρείτε ότι αυτό θα το δει η κοινή γνώμη. Θεωρείτε ότι θα είστε κάποιος που θα μπορεί να εμπιστευθεί ο μέσος πολίτης να είναι αυστηρότατος κριτής και ελεγκτής. Συνάδελφοι, εντάξει το ξέρω ότι είναι ακρόαση, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γίνει ανάκριση, δεν χρειάζεται να απαντήσει με τέτοιο τρόπο τώρα η, η υποψήφια. Ε, Τίθεται θέματα ερεύνησης συνείδησης. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση αυτή. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωριζόμαστε εδώ και καιρό και από την Ολομέλεια. Δεν είναι καθόλου απλή, ούτε εύκολη ήταν η απόφαση τώρα πραγματικά να αλλάξω ε, καριέρα και να ε, φύγω από την πολιτική αλλά δεν είναι κάτι το ξένο ε, για μένα. Ε, θα ήθελα να το επαναλάβω. Το έχω ξανακάνει αυτό και το έχω γράψει. Ήμουν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και ανέκαθεν ε, προσπαθούσα να εργάζομαι με αντικειμενικότητα, με αμεροληψία, με τρόπο αδέκαστο και ανεξάρτητο. Και πάντα υπήρχαν συγκρούσεις συμφερόντων. Το θέμα δεν είναι να τις αποφεύγει κανείς, αλλά ε, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με συγκρούσεις συμφερόντων θα πρέπει να μπορεί ο καθένας και εγώ προσωπικά να υπερασπίζω την ε, άποψή μου. η θητεία του Ευρωβουλευτή είναι κάτι που έχει πεπερασμένη ε, ισχύ και μετά ε, θα ακολουθήσω όλα αυτά που ορίζει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου, ε, κανονισμοί της Όλαφ και του Ελεκτικού Συνεδρίου και τα λοιπά και θα ανταποκριθώ στο ρόλο και στο καθήκον μου. Ο καθένας έχει την προσωπική του γνώμη, την ιδιωτική γνώμη. Αυτό ισχύει και μέσα σε ένα πολιτικό κόμμα και μέσα σε μια πολιτική ομάδα. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάντα τις ίδιες απόψεις. Ούτε πρόκειται τώρα να απαριθμίσω όλες τις περιπτώσεις όπου διαφώνησα με την πλειοψηφία της ομάδας μου ή ε, του κόμματος. Αλλά κάθε φορά που έπαιρνε κατά πλειοψηφία μία απόφαση η πολιτική μου ομάδα, εγώ ήμουν υποχρεωμένη να τη σέβομαι και να την υποστηρίζω και να μην την αφισβητώ, ακόμα και αν διαφωνούσα. Ακόμα και αν θεωρούσα ότι δεν ταυτίζεται 100% με τις προσωπικές μου απόψεις αποφάσεις. Μην ανησυχείτε. Μήπως θεωρήσει κανείς στην Ουγγαρία ότι είμαι πολιτικός έτσι ανερμάτιστη. Ο κόσμος στην Ουγγαρία θεωρεί ότι είμαι ειδικό. Ε, έχω περάσει από το πανεπιστήμιο, προέρχομαι από το πανεπιστήμιο Υπάρχουν ε, πολιτικοί που αρέσκονται στο να συζητούν θέματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα. Αλλά εγώ μπορεί να είμαι πολιτικός, αλλά μιλώ για θέματα τα οποία γνωρίζω. Και όταν δεν τα γνωρίζω, ε, το αφήνω συναδέλφους που είναι σοφότεροι από μένα. Έχω άλλους δύο συναδέλφους και παρακαλώ να περιοριστείτε στο ένα λεπτό έκαστο. Και θα τα ομοδοποιήσουμε. Ο κύριο Αλαφράγκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι συμφωνώ με την κυρία, μάλλον ε, ήμασταν με την κυρία Γκάλ Πέλτσε στην ίδια πολιτική ομάδα, αλλά δεν είχα και ποτέ τη δυνατότητα να συνομιλήσω μαζί της ε, ε, και τώρα τη βλέπω και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνω πως ε, έχει ένα βιογραφικό σημείωμα που είναι πολύ δεδειγμένο σε σχέση με το αντικείμενό της. Ε, είναι ελέγκτρια, έχει εκπαιδευτεί στα φοροτεχνικά ζητήματα, ήταν εδώ ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, έχει ασχοληθεί με τα χρηματοπιστωτικά. Στις γραπές της απαντήσεις βλέπω ότι έχει να κάνει περισσότερο με αναθεώρηση λογαριασμού με Ευρωπαϊκή ε, τράπεζα, Τραπεζική Αρχή, Ασφάλεια, Συντάξει κτλ. Δεν είναι κατά την άποψή μου τόσο θέμα πολιτικής, ε, το που ανήκει πολιτικά κάποιος, αλλά αυτή ε, οι δυνατότητες, έχει τι ικανότητες ε, και από την διασταδιοδρομία βλέπουμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνάδελφο ότι το έργο της πραγματικά είναι εξωσέβαστο εδώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι το να είναι κανείς ευρωβουλευτής ε, είναι για να είναι κανείς μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν θα είστε ούτε πρώτη τελευταία. Ε, ο πρόεδρος, ο πολύ σημαντικός πρόεδρος τώρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διατέλεσε ευρωβουλευτής και υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Ο κύριος Φάμπρα Βαγιές, δικός μου ε, συμπατριώτης, δυστυχώς απεβίωσε, ήταν μέλος και αυτής της Επιτροπής. Θέλω να σας ρωτήσω, διάβασα το ερωτηματολόγιο και σε σχέση και με τις ερωτήσεις που κατέθεσαν άλλοι στην άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, η σχέση μεταξύ αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και του Ελληνικού Συνεδρίου, η αμεσότητα, η ταχύτητα των εκθέσεων, τι μπορούμε να πούμε ε, θα περνάνε λίγο πιο γρήγορο στην εκπόνηση των εκθέσεων το Ελληνικού Συνέδριου. Αυτή είναι η άποψή μα. Και δεύτερον, η συνεργασία με τι Εθνικέ Ελεγκτικέ Αρχέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει από τι Εθνικέ Αρχέ μεγάλο τμήμα των ε, στοιχείων. Πώ το βλέπετε εσεί και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την συλλογή δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Deutsch, bitte. Ο κύριος Ντόιτς παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, θα συνεχίσω πιάνοντας το θέμα από εκεί που τάφησε ο κύριος Αλαφράγκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέλη του Ελεκτικού Συνδρίου να εργάζονται με επαγγελματισμό. Να είναι απολύτως ανεξάρτητη. Όπως είναι επίσης η απέτηση για οποιονδήποτε ελεγκτή, έτσι ισχύει και για αυτούς που διατέλεσαν κατά παρελθόν ευρωβουλευτές. Έχουμε δει ε, τα αποτελέσματα από το Βούλγαρο, τον Φιλανδό ελεγκτή και το Γερμανό συνάδελφο. που ήταν κατά παρελθόν ευρωβουλευτές, πολιτικοί και οι τρεις. Άρα δεν νομίζω ότι και στην προκειμένη περίπτωση θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εξάλλου, τα ικανότητα, τα ικανότητες, τα προσόντα σας ε, είναι αξιοσημείωτα, ε, είναι δειγμένα. και Γκάλ Πέλτς, ε, επίσης έχει φροντίσει πολύ συχνά και έχει δείξει ότι είναι ανεξάρτητη κατά το έργο της και στις ε, ψηφοφορίες. Έδειξε ότι είναι αμερόληπτη και τη στήριξαν και διάφορες πολιτικές ομάδες. Υπήρξε και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αμφιβολία. Βέβαια υπάρχει το εξή θέμα. Υποψήφια. Μπορεί να βοηθήσει για να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Ελεκτικού Συνεδρίου, ώστε να μπορούν από κοινού ε, τα δεύτερα θεσμικά όργανα να φροντίσουν να σταματήσει τα παιχνιδάκια που παίζει το Συμβούλιο. στην απαλλαγή και σε άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με τον προπολογισμό ε, δεν ε, αντιμετωπίζει ως εταίρο τα άλλα διθεσμικά όργανα το Συμβούλιο. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρει έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Γι' αυτό και η σχέση μας ε, είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι και εγώ που η συνάδελφος είναι γυναίκα. Αλλιώς. Ε, δεν θα μπορούσε να απαντήσει με τον τρόπο που απαντά από τις αηδίες που τις ε, προσάπτουν οι ε, αριστεροί εδώ στο Κοινοβούλιο. Μιλήσαμε για την έκτακτη έκθεση. Δεν θέλω να μιλήσω για ένα ποσό ε, και για την πληθώρα των ειδικών εκθέσεων ε, οι οποίες συζητώνται και διεκπεραιώνονται και μετά εξαφανίζονται. Δεν θα μπορούσε το ελεγκτικό συνέδριο να προβληματιστεί τι θα γίνει με τις ειδικέ εκθέσεις και τι συνέχεια πρέπει να δίνεται μετά τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας. Δεύτερον, και στις κανονικές εντός εισαγωγικών εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου υπάρχουν κάποιες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συζητάμε λίγο και μετά αυτό εξαφανίζεται στο γενικότερο χάος στην Ιρβάνα κάπου. Καλό θα ήταν να δίνεται συνέχεια και σε αυτό και να έχουμε και πληροφόρηση ε, το Κοινοβούλιο για το τι απέγινε αυτή η έκθεση. Και ένα τρίτο, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών και με το Κοινοβούλιο, νομίζω θα μπορούσε να ενισχυθεί από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου. Γιατί ειδικά στην Επιτροπή μας εδώ ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ ε, αυτά που επεξεργαζόμαστε να ε, έχουν συνέχεια και όχι μια βραχία ζωή και μετά να σκάνε, να εξαφανίζονται. Ο Πολωνός υποψήφιος καταψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο, παρόλα αυτά όμως τον επιβεβαίωσε ε, το Συμβούλιο. Εσείς πώς θέλετε να συνεργαστείτε στο μέλλον ως πρώην Ευρωβουλευτής και με αυτόν τον συνάδελφο. Ο κύριος Φλάναγκαν για ένα λεπτό. Είπατε ότι θέλετε να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα των γυναικών. Ο ηγέτης του κόμματός σας, το οποίο θέλετε από ό,τι φαίνεται να παραμείνετε μέλος, δεν είναι και πάρα πολύ υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Ούτε καν στη συμμετοχή των γυναικών στην ουγγρική πολιτική. γιατί λέει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αντέξουν και να ανεχθούν τη συνεχή δολοφονία χαρακτήρων. Ελπίζω εσείς να έχετε έτσι αρκετό τσαγανό. Πού συμφωνείτε με τον πρόεδρό σας και εκεί που διαφωνείτε του τα έχετε πει, γιατί σε τελική ανάληξη πρέπει να δείξετε χαρακτήρα. Αυτή η δουλειά αυτό θέλει. Και εγώ ε, ε, έχω ε, πραγματικά τρομοκρατηθεί. Έχουμε εδώ βουλευτή που θεωρεί ότι ε, ε, είναι τέλειο το βιογραφικό σας. Αν είχε πάει κάποιος από τη δική μου οικογένεια στη χώρα σας, θα τον είχατε εκδιώξει. Τι γίνεται με τις γυναίκες πρόσφυγες. Οι μετανάστες θα μπορούν να δουλεύουν. Οι πρόσφυγες που προσπαθήσετε να εκδιώξετε από τη χώρα σας, επιτρέπετε να δουλεύουν. Τα έχετε πει αυτά στον ηγέτη σας γιατί δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στο κόμμα σα. Κύριε Φλάνακαν, η ερώτησή σας δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συζητούμε τώρα εδώ. Εγώ πιστεύω ότι έχει. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Έχετε δείξει χαρακτήρα απέναντι στον ηγέτη σας με τις ρατσιστικές απόψεις. Ε, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Την έχετε ε, κάνει την ερώτηση. Δεν μου απάντησε εάν έχει βρεθεί απέναντι στον ηγέτη της. Και, και δεν με υποστηρίζει κανείς. Κοιτάξτε, δεν θα συζητήσουμε το ΦΙΤΕΣ. Εγώ δεν θέλω να είμαι ούτε μέλος του ΦΙΤΕΣ, ούτε μέλος της οικογένειάς σας. Το τι προτιμάει ο καθένας εδώ πέρα μέσα δεν είναι θέμα συζήτησης αυτό που είναι για μένα σημαντικό να είμαστε δίκαιοι απέναντι σε όλους τους υποψηφίους και σωστοί. Δεν είναι σωστή αυτή η ερώτηση, αυτές οι ερωτήσεις. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ερώτηση σε υποψήφιο που συμφωνείς με τον αρχηγό του κόμματό σου και που όχι. Δεν είναι αντικείμενο της συζήτησης. Κοιτάξτε, εγώ προεδρεύω εδώ. Λοιπόν, και το λέω. Και σε εσά ως μέλος, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρούμε κάποιες διδικασίες εδώ. Είμαι πάρα πολύ βεπισμένη ότι μπορεί και να, να απαντήσει. Έχει απάντηση και σε αυτό η υποψήφια. έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις. Και φυσικά και θα απαντήσω και στις ερωτήσεις του κυρίου Φλάναγκαν. Και το επιτρέπει η κυρία Σμιτ, θα περάσω σε αυτή την ερώτηση του κυρίου Φλάναγκαν. Εδώ και 10 χρόνια είμαι η μόνη γυναίκα που είμαι στο Προεδρείο ε, του Φίντες και μπορεί αυτό να μην είναι τίποτα. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι περιφρονεί, ίσως και μισεί ο αρχηγός του κόμματος, τις γυναίκες μέλη του κόμματος. Ε, τέλος πάντων, ε, αφήστε με να πω κάτι βουλευτής ε, στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη, αλλά έχω εγώ το λόγο τώρα. Συζητήσαμε το θέμα της ποσόστοσης γυναικών, υπήρξε μια πάρα πολύ τόνη συζήτηση και ξέρετε ποιος με στήριξε και ποιος στήριξε τις δικές μου απόψεις. Ο αρχηγός του κόμματός μας. Γι' αυτό τις ποσοστώσεις των γυναικών. Βέβαια η ψηφοφορία δεν ήταν επιτυχή στο τέλος, αλλά όταν ήρθα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελα να το θέσω και, αυτό το, και εδώ το θέμα αυτό προς συζήτηση. Ξεκίνησα πολύ νωρίς, δεν είχα καμία υποστήριξη και στο ΦΙΝΤΙΣ και στο Αγγλικό Κοινοβούλιο δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό το θέμα των ποσοστώσεων, αλλά εγώ δεν θα εγκαταλείψω τις προσπάθειές μου. Θα το ξαναπροσπαθήσω αν μου δοθεί ευκαιρία και στο πλαίσιο της οικογενειακής πολιτικής προσπάθησα να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα, δηλαδή να έχουν περισσότερες γυναίκε σε υψηλά αξιώματα, σε ηγετικέ θέσεις, να υπάρχει καλύτερη συμφιλίωση επαγγελματικού, οικογενειακού βίου και ε, μεγαλύτερη ισότητα και τα λοιπά, μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις γυναίκες, για να προχωρήσουμε. Τώρα για το επαγγελματική μου σταδιοδρόμιο και το βιογραφικό μου, τα μελετήσατε ε, και τα είπα όλα και εδώ πλέον τα έχετε υπόψη. Ναι. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις ε, στο κόμμα μας. Το ΦΙΔΕΣ φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και σε εσά, παρ' όλα αυτά ανήκετε σε ένα κόμμα όπως και εγώ ανήκω σε ένα κόμμα, στο δικό μου κόμμα. Και διαφωνώ για πολλά ζητήματα. Έχω άλλες απόψεις, δεν, μπορώ, δεν θέλω να σας αναφέρω συγκεκριμένα τώρα. Ε, στη συνδέωση του Προεδρείου του Κόμματος που εγώ ε, έχω διατυπώσει διαφορετικές απόψεις σε ποια θέματα. Πιστέψτε με απλά ε, ότι ως γυναίκα μπορώ να έχω για συγκεκριμένα στήματα διαφορετική άποψη. Έρχομαι στον κύριο Σάλα Φράγκα και θέλω να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια, για την επαγγελματική εμπειρία, την αμυγός επαγγελματική εμπειρία Πράγματι είμαστε βουλευτέ, είμαστε και στην ίδια πολιτική ομάδα, αλλά το σημαντικό είναι ότι μπορεί να μην γνωρίζουμε όλοι ε, την ε, παρελθούσα εργασιακή εμπειρία, τι έχει κάνει ο καθένας. Εργαζόμαστε απλά εδώ πολύ σκληρά για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον ε, για τα παιδιά μας. Και αυτό είναι το σημαντικότερο σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδρου και των Εθνικών. Σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν πολύ τα πράγματα. Δεν έχω ε, εγώ προσωπικά έντονη συμμετοχή σε αυτή τη σχέση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, συμμετέχουν και να ε, ενσωματωθούν πολύ περισσότερες εργασίες εργασίε του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου οι εθνικέ ελεγκτικέ αρχέ για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όμω αυτό που δημιουργεί ένα πρόβλημα εδώ είναι το περιεχόμενο των πληροφοριών και η μεθοδολογία. Εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε μια προσέγγιση ε, σφαιρική, συνολική. Τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια πιστεύω ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν περισσότερα καθήκοντα ε, και να έχουν ένα μεγαλύτερο ρόλο στο πλαίσιο των ελέγχων. Ένα άλλο σημείο, για το οποίο δεν δέχτηκα πολλές ερωτήσεις. Είναι το λεγόμενο DAS, ε, δήλωση εξοπιστίας. Δεν έχει συζητηθεί πολύ αυτό το θέμα. Είναι πολύ δύσκολο με έναν και μόνο δείκτη και με μία και μόνο δήλωση να αξιολογήσουμε και να συνθέσουμε τα αποτελέσματα πολλών ετών. Θα μπορούσε ίσως να γίνεται ε, στη μέση της χρονιάς ή μετά από κάποια μετά άλλη προθεσμία να ξαναγίνεται αυτός ο έλεγχος. Τώρα για τον κύριο Deutsch πράγματι 6-7 χρόνια, ίσως και περισσότερο, είχαμε δει την ε, στάση του Συμβουλίου, που πραγματικά δεν ε, στέκεται στο πλευρό μας πολλές φορές. Υπάρχουν πάντα δύο νομίσματος βέβαια. μπορεί το Συμβούλιο να επικαλείται ένα πρωτόκολλο υπεραρχαίο από το 1970 που μιλά για τη συνεργασία των θεσμικών οργάνων κτλ. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για την υλοποίηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής. Και πραγματικά είναι πολύ κακό το μήνυμα ε, το οποίο εκπέμπει το Συμβούλιο ότι όλοι οι άλλοι θεσμοί και ο διαμεσολαβητής και τα λοιπά να απαντούν ε, όλες τις ερωτήσεις και μόνο το Συμβούλιο να μην ε, λογοδοτεί απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν, κακό, δεν είναι καλό αυτό. το να βάζει ε, στην ιστοσελίδα του το Συμβούλιο μόνο κάποιες απόψεις δεν δείχνει ότι θέλει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και δεν, όταν δείχνει ότι δεν θέλει να απαντήσει σε ερωτήσεις τους των Ευρωβουλευτών για την κυρία Σμιτ, ε, για τις ειδικέ εκθέσεις, ότι πρέπει κάτι να γίνει. Ναι, πράγματι, πρέπει να εστιάσουμε, πιστεύω, σε θεματικούς τομείς. Δεν έχουμε πολλούς πόρους, είναι πολύ περιορισμένοι πόροι. και διάθεση των πόρων ένα δημιουργεί πρόβλημα. Σίγουρα και δεν είναι καλό τα αποτελέσματα των ειδικών εκθέσεων κάπως να ε, εξαφανίζονται, να μπαίνουν σε ένα σιρτάρι. Φυσικά έχουμε δαπανίσει ανθρώπινους πόρους ε, και υλικούς πόρους και μετά δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Άρα ποια είναι η λειτουργία και η χρησιμότητα αυτών των ειδικών εκθέσεων αν δεν έχουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα και αν παραμένουν οι συστάσεις μόνο στα λόγια και αν το περιεχόμενο των ειδικών εκθέσεων δεν συζητείται. Άρα δεν μπορούν να ακολουθήσουν ή να προκύψουν από τις συστάσεις αυτές κάποιες νομοθετικές προτάσεις. Και στην κατάρτιση του προπολογισμού και του δημοσιομικού σχεδιασμού. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικές εκθέσει, γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να πετύχουμε του στόχου μας. Μπορούμε να πούμε ναι, ωραία, τα αποτελέσματα, ο λογιστικός έλεγχος και το ένα και το άλλο. Πρέπει να υπάρχει μια διασταύρωση και μια διασύνδεση. Νομίζω ότι απάντησα όλες ε, τις ερωτήσεις. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος Σάκ που δεν τον είχα δει μέχρι τώρα. Ναι, πρόεδρε. Είχα σηκώσει το χέρι μου, αλλά δεν είχα καταλάβει αν με είχατε δει. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Το ελεγκτικό συνέδριο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παράλληλα, ο Όλαφ είναι και αυτός συναρμόδιος για την καταγγελία κάποιων παραβάσεων ή και απάτης. Να υπογραμμίσω επίσης ότι το ελεγκτικό συνέδριο συνυπέγραψε την διαθεσμική συμφωνία που δίδει αρμοδιότητα στον Όλαφ για να διεξάγει έρευνες και επί του ελεγκτικού συνέδριου. και επί τη βάση των ερευνών του Όλαφ θα πρέπει να παραπεμφθεί ένα μέλος του ελεκτικού συνεδρίου και βρίσκουμε λοιπόν μπροστά μας ένα παράδοξο. Ο Όλαφ ελέγχει κάποιες δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων εκείνων και των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου, ενώ παραλλήλως και παραδόξως το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσε να διεξαγάγει έρευνες επί των δραστηριοτήτων του Όλαφ. Την ίδια στιγμή. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για αυτή την κατάσταση που είναι ε, λίγο περίπλοκη δομή και παράδοξη. Και θα ήθελα να καταλάβω αν θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική αυτή η κατάσταση για τη διάκριση των εξουσιών. Απάντηση. Βεβαίω κάθε σύστημα έχει τα υπέρ και τα κατά του και ελλείψεις φυσικά. Τα κατά και οι ελλείψεις φαίνονται κατά τη λειτουργία ενός συστήματος. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά γύρω μας. Έχουν αλλάξει και λογιστική ελέγχοι. Την τελευταία επταετία το ελεγκτικό συνέδριο έχει αποκτήσει νέες εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Το γεγονός ότι διεξάγονται έρευνες κατά μελών του ελεγκτικού συνεδρίου ισχύει. Τώρα αν είναι αυτό κάτι παράδοξο και περίπλοκο, δεν το ξέρω. Βεβαίως θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει σωστά τη δουλειά του και να ελέγχει και τον προϋπολογισμό της Όλαφ, εάν γίνεται σωστά η εκτέλεση και νομότυπα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Είναι σωστό. Το παράδοξο που περιγράψατε εσείς φυσικά πρέπει να λυθεί και υπάρχει διοργανική συμφωνία μεταξύ Όλαφ και Ελεκτικού Συνεδρίου για τους τομείς εκείνους που μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Και φυσικά τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου όταν βλέπουν ε, ότι υπάρχει μια τετασταλία, μια παρατυπία ακόμα και απάτη, οφείλουν να προβαίνουν στα απαραίτητα βήματα και στις απαραίτητες ενέργειες. Ακόμα και αν αυτό αφορά την Όλαφ. Βεβαίως πάντα χωράνε βελτιώσεις Αλλά όλα λύνονται με τη συνεργασία και με τη συζήτηση. Και βέβαια θα πρέπει να αξιοποιούμε και τις εμπειρίες μας για να βελτιώνουμε πάντα το νομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής για να κλείσει. Κύριε Τάραντ, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πάντοτε Ήμουν θαυμαστή του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται τι εργασίε τη Επιτροπής, διευθύνεται μάλλον. Και παρότι έχετε δίκαιο ότι τα ερωτήματα του κυρίου Φλάναγκαν πήγαν πέραν της θεματικής του ελέγχου και του ελεκτικού συνεδρίου, κατά την άποψή μου τα μέλη πρέπει να έχουν το λόγο να υποβάλουν οποιασδήποτε ερωτήσεις επιθυμούν, διότι εδώ εκπροσωπούμε διάφορους πολίτες, διάφορους ψηφοφόρους. Τώρα εγώ υποτίθεται ότι πρέπει να συντάξω μια έκθεση, επί της οποίας θα ψηφίσουμε. Και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, διότι περπατάω σε λεπτό πάγο όπως είπε ο κύριος Φλάναγκαν, δεν είναι όλοι οι μετανάστες κακοί άνθρωποι και ούτε όμως όλα τα μέλη του Φίντες. Και η πορτένη αυτή νομίζω ότι μάθαμε πολλά για τις θέσεις και τις απόψεις της κυρίας Γκάλ Πέλς και σκέπτομαι να συντάξω μια θετική έκθεση. Διατηρώντας υπόψη όμως ότι πρέπει να προωθήσουμε το θέμα των συνθήκων. Γιατί προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση όλα αυτά δεν ε, βλάπτουν το Συμβούλιο. Δηλαδή, οποιαδήποτε και να είναι η τελική μας απόφαση δεν θα πρέπει ε, το Συμβούλιο να μπορεί να την αλλάξει. Μάλιστα. Ε, εδώ τελειώνει η δημόσια ακρόαση. Επιθυμούν οι πολιτικές ομάδες να συνεννοηθούν Παρακαλώ όσους δεν ψηφίζουν και είναι σύμβουλοι πάλι πολιτικών ομάδων να αποχωρήσουν για ένα τέταρτο το πολύ. Μάλλον όσοι δεν είναι μέλη ή υπάλληλοι και σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων, όλοι οι άλλοι να αποχωρήσουν. Μυστική ψηφοφορία θα ακολουθήσει. Μικρή διακοπή για τις πολιτικές ομάδες για πέντε λεπτά και κάτι. 11 παρα θα ξαναρχίσουμε. Και Σας παρακαλώ όλοι οι υπόλοιποι να αποχωρήσετε. Όσοι δεν δικαιούστε να παραμείνετε κατά τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης μας που θα γίνει και κλεισμένα των θύρων για την ψηφοφορία.